Ιδιαίτερα ικανοποιητικό είναι το ότι 35% των βουλευτών είναι γυναίκες, το υψηλότερο ποσοστό μέχρι σήμερα. ...170 εκατομμύρια πολίτες ψήφισαν στις εκλογές και η δική μας δουλειά αγαπητοί συνάδελφοι εξυπηρετεί ένα μεγάλο στόχο την ένωση της υπήρου, της υπήρου μας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ κατά τη διάρκεια των εργασιών μας πως βασιζόμαστε σε κάποιες αξίες, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ελευθερία, τη δημοκρατία, το δικαίωμα στην ειρήνη. Αυτές είναι οι βάσεις των όσων κάνουμε. Μας συνδέει η αλληλεγγύη. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω αγαπητοί συνάδελφοι πάντα να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Εάν συμβαίνει αυτό, θα είμαστε και επιτυχείς. Θα ήθελα να περάσουμε τώρα στο έργο της σημερινής ημέρας. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω πως σύμφωνα με τον κανονισμό υπό την προεδρία του αποχωρούντος Προέδρου δεν μπορεί να γίνει καμία άλλη συζήτηση παρά μόνο η εκλογή του Προέδρου και η εξέταση των εντολών. Σας ανακοινώνω πως έχουν σχηματιστεί οι εξής κοινοβουλευτικές ομάδες. Η ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, οι Χριστιανοδημοκράτες, ΕΛΚ, η ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η κοινοβουλευτική ομάδα της ε, Συμμαχίας